Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Επειδή ήδη έχουμε κάποια καθυστέρηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή τη συνεδρίαση. Θα πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ας την εγκρίνουμε. Δεν έχω καν ανακοινώσει του Προέδρου, οπότε Μπορούμε αμέσω να περάσουμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη και να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο Όλιβερ Φαρχέλη που θα μα παρουσιάσει τι φρέσκε μόλι βγήκαν από το φούρνο, προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό τη μεθοδολογίας για τη διεύρυνση. Κύριε Επίτροπε, ε, εκτιμούμε ιδιαίτερω που ήρθατε για την ανταλλαγή απόψεων, γιατί ευθυγραμμίζεται η προθυμία σας με την ε, εδρεωμένη πλέον πρακτική της υποβολής σημαντικών προτάσεων πρώτα και απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να γίνεται πλήρω σεβαστό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μπορούν και οι ευρωβουλευτέ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και τον έλεγχο τη ενταξιακή διαδικασία. Μια και έχουμε μόνο τρία τέταρτα στη διάθεσή μα, θα σα θέρμο παρακαλούσα να περιοριστείτε στην εισαγωγική σα ομιλία σε 10 με 12 λεπτά το πολύ για να έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Επίση, θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου ομιλία των Ευρωβουλευτών. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και την οργάνωση αυτή τη έκτακτη συνεδρίαση ε, για να σας παρουσιάσω τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεθοδολογία της διεύρυνσης ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία μου εδώ, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, για να σας παρουσιάσω τα σχέδιά μας για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η, Ευρωπαϊ... η διαδικασία της διεύρυνσης είναι ύψητη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε μια αξιοκρατική ενταξιακή διαδικασία που είναι προς το οικονομικό φελός μας αλλά και για την ασφάλεια και η γεωστρατηγική μας επένδυση σε μια σταθερή και ισχυρή εύρωστη ενωμένη Ευρώπη. Τρεις είναι οι άξονες ε, των εργασιών μας και έτσι προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την διαδικασία της διεύρυνσης. Πρώτον, θα αναθεωρήσουμε τη μεθοδολογία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Στη συνέχεια θα έχουμε τον δεύτερο άξονα με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Και τρίτον, οι οικονομικές αναπτύξεις και σχέδιο επενδυτικό για το σύνολο της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, που θα υποβάλουμε στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ που θα γίνει 6 και 7 Μαΐου. Η πρότασή μας για την αναθεωρημένη διαδικασία διεύρυνσης θα καταστήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ε, πιο αξιόπιστες, πιο προβλέψιμες, πιο δυναμικές και ε, υπό ισχυρό πολιτικό πηδάλιο. Ε, έχουμε αναθεωρήσει και ουσιαστικά ενισχύσει τη διαδικασία. Αλλά βασικό στόχος είναι η διεύρυνση, η ένταξη, συγγνώμη, ε, πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα εργαλεία και, το μηχαν... και τους μηχανισμούς μας, ώστε οι εταίροι μας, χάρη στην οικονομία και το κράτος δικαίου, να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι σχετικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν πραγματικές συνέπειες, να προωθούν την ευημερία, να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο και να δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας στις χώρες και στους λαούς της περιοχής. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων παραμείνει όχι μόνο δυναμικός αλλά και επιταχυνθεί ταυτόχρονα. Και η πρόταση για μια αναθεωρημένη μεθοδολογία εδράζεται σε τέσσερις αρχές. Αρχή πρώτη, αξιοπιστία. Η ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να εδράζεται σε μια ε, σταθερή εμπιστοσύνη και αμοιβαία επίσης εμπιστοσύνη. Και μάλιστα η οι ηγέτε των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι στι μεταρρυθμίσει που απαιτούνται, ιδιαίτερα στο κράτο δικαίου, για να καθησυχάσουν ε, τις εύλογες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών χωρών. Και επίσης ε, θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στις θεμελιώδεις ελευθερίες που είναι ο πυρήνας της πραγματικής αλλαγής. Κράτος δικαίου, δημοκρατία, θεσμι... Ε, δημοκρατικοί θεσμοί και οικονομικά κριτήρια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει την υπόσχεση για μια αξιοκρατική προσέγγιση όταν οι χώρε εταίροι εκπληρώσουν τα απαραίτητα κριτήρια, θα πρέπει να περνάνε στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Δεύτερη αρχή, ισχυρό πολιτικό πιδάλιο. Δεδομένη τη πολιτική φύση τη διεύρυνση, η διαδικασία θα πρέπει να τύχει μια ε, ισχυρή πολιτική καθοδήγηση και από τι δύο πλευρέ. Θέλουμε σημαντική δέσμευση των υποψηφίων χωρών μέσω τακτικών συνόδων κορυφής, αλλά και υπουργικών διασκέψεων. Επίσης, θέλουμε να εμπλέξουμε περισσότερα τα κράτη-μέλη και να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθούν και να επανεξετάζουν τη διαδικασία, να στηρίζουν και να παρακολουθούν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Επίσης, τρίτη αρχή, μια πιο δυναμική διαδικασία. Για να ενισχύσουμε το δυναμισμό, θα ομαδοποιήσουμε τα κεφάλαια της διαπραγματεύση σε έξι θέματα. Θεμελιώδεις αρχές, ανταγωνιστικότητα, ε, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βιώσιμη συνδεσιμότητα μαζί με την γεωργία, πόρους και διαπραγματεύσεις. Επίσης, ε, θέλουμε πιο πολιτικές συζητήσεις στις θεματικές ενότητες, προκειμένου να έχουμε από την αρχή ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε, η διαπραγματεύση για κάθε θεματική οντότητα θα ξεκινούν για το σύνολο των κεφαλαίων. Επίση, θα θεμελιώδη δικαιώματα, κράτο δικαίου, οικονομικά κριτήρια και μεταρρύθμιση τη δημόσια διοίκηση, αυτό το κεφάλαιο, αυτή η θεματική οντότητα θα είναι αυτή που θα, θα αρχίζει πρώτη και θα ολοκληρώνεται τελευταία. Γιατί θα πρέπει μεταρρυθμίσει να προηγηθούν σε αυτή τη θεματική ενότητα πριν ξεκινήσουν άλλε ή πριν αρχίσουν άλλε ανοίξουν άλλε για διαπραγματεύσεις. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της θεματικής ενότητας και το κλείσιμο του κεφαλαίου θα πρέπει να είναι το πολύ ε, ένας χρόνος κατά προτίμηση. Επίσης θέλουμε προβλεψιμότητα και για τις δύο πλευρές. είναι από το τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ε, υποψήφιες χώρες, καλύτερος προσδιορισμός των προϋποθέσεων και το θετικό αντίκτυπο σε περίπτωση επιτέλους πρόοδου και αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση ε, μη επίτευξη πρόοδου. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι σαφή. Επίσης να δώσουμε ενάυσματα εφόσον εφαρμόζονται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να έχουμε σταθερή, σταδιακή ένταξη στις πολιτικές της αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσο ταχύτερες είναι οι μεταρρυθμίσεις, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει το, στην ενταξιακή της πορεία η χώρα. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει παρατεταμένη στασιμότητα ή παλινδρόμηση. Και Επίσης θα πρέπει να έχουμε πιο αποφασιστικά μέτρα που θα διορθώνουν την περίπτωση σε περίπτωση παλιδρόμησης στασιμότητας. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στη σύστασή τη για την έναρξη συνταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Και ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσουν αυτέ πριν τη Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ το Μάιο. Γιατί και οι δύο χώρε έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια και έχουν κάνει τι μεταρρυθμιστικέ του προσπάθειε. Βέβαια, παρακολουθούμε την πρόοδό του και θα ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη ε, ω ονούπο κατά πάσα πιθανότητα στη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Γιατί για να στα αξιόπιστη εταίροι πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Και προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ θα καταθέσουμε και προτάσεις ε, με ιδιαίτερο επίκεντρο την οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να, να κάνουμε πιο αισθητή την παρουσία μας στα Δυτικά Βαλκάνια, να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας και να γεφυρώσουμε το οικονομικό χάσμα μεταξύ ημών και των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, όπω βλέπετε, και θα χρειαστούμε την υποστήριξή σα για να το υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε από κοινού τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να προωθήσουμε τι επενδύσει στα Δυτικά Βαλκάνια και να στηρίξουμε την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των χωρών αυτών για καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα και να αποφύγουμε τη διαρροή εγκεφάλων και ταλέντων από την περιοχή. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Επίτροπε Βαρέη, σας ευχαριστούμε για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Έχουμε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν θα τα καταφέρουμε να δώσουμε σε όλους το λόγο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τους συντονιστές. Δύο λεπτά στον καθένα εκ μέρους του ΕΛΚ ο Μιχαήλ Γκάλερ. Ευχαριστώ Επίτροπε και σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε την ανακοίνωση αυτή εδώ απευθείας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς ως ε, ΕΛΚ χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε την ανακοίνωση αυτή για την ε, νέα στρατηγική για τη διεύρυνση. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αναζωογονείται αυτή η διαδικασία, όπου ενισχύεται η αξιοπιστία μας και ενισχύεται ο πολιτικός χαρακτήρας της διαδικασίας. Με την θέσπιση κριτηρίων για τους υποψήφιους θεωρούμε ότι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αυτή και έτσι γινόμαστε και αξιόπιστοι και απέναντι στα υπάρχοντα κράτη-μέλη ότι ε, παραμένουμε σε μια διαδικασία όπου αν υπάρξει οπισθοδρόμηση θα μπορέσουμε να ε, ανέρεσουμε ή να μπλοκάρουμε ε, κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί. Είναι θετικό το ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουμε χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξη σε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία υπάρχουν για τα κράτη-μέλη κάτι που επίσης ε, θα λειτουργήσει ενισχυτικά. Πολιτικά, επίσης, θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί που θα συμπεριλαμβάνουν, θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κρατών μελών στις διαπραγματεύσεις με εμπειρογνώμονες, ώστε να ενισχυθεί η αφοσίωσή τους, η προσήλωσή τους και η συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία και να μην γίνεται όλο αυτό το πράγμα μόνο μέσα από, από τις Βρυξέλλες. Ελπίζουμε στη διαδικασία να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαιρετίζω ιδίω το γεγονό ότι δίνεται προσοχή και μεγάλη έμφαση στην, ε, στο κράτος δικαίου, στην παρακολούθηση και ένας ε, πιο ισχυρός πολιτικός ρόλος για τα θεσμικά μας όργανα. Ευχαριστούμε Μίχαελ Γκάλα. Πρωτού δούμε το βιντεάκι στην οθόνη. Θα δώσω το λόγο στον τον Νίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ. αξιότιμο Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωσή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και χαιρετίζουμε τη νέα προτινόμενη μεθοδολογία για την προσχώρηση. Η ευρωπαϊκή ιστορία είναι ιστορία διεύρυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανανεωθεί εξωτερικά-εξωτερικά ταυτόχρονα. Καθώ η μία διαδικασία δεν αποκλείει την άλλη. Είναι θετικό το γεγονό ότι η Κομισιόν επαναλαμβάνει την ε, ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, κάτι που εμεί, οι Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζαμε πάντοτε. Και θέλουμε την πλήρη αφοσίωση και προσήλωση της Κομισιόν στην διαδικασία διεύρυνσης. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την ανακοίνωση η οποία συμπεριλαμβάνει τη δήλωση ότι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί προτεραιότητα. Κάποια ερωτήματα. Ο μόνιμο ως μόνιμος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μαυροβούνιο θέλω να πω το εξής. Αν η μεθοδολογία ε, ε, αφορά και τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ή μόνο τις χώρες για τις οποίες πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία διεύνησης. Στην δήλωση του Συμβουλίου αναφέρεται ότι θα είναι δική του επιλογή. Θέλω να μάθω ε, σε αυτή την περίπτωση των δύο χωρών τι θα γίνει. Υπάρχει ήδη κάποιο σχέδιο για αυτές τις χώρες, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν κάποια αρχικά σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν. Για για την αντιστρεψιμότητα. Εσείς ε, ε αναφερθήκατε σε αυτήν ότι μπορεί να γίνει μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε έξι χρόνια, σε χρόνια σκοπεύετε να ολοκληρώσετε αυτές τις μακροχρόνιες ε, και επίπονες διαπραγματεύσεις. Για το Renew, η κυρία Βάουτμαν, έχει το λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ναι, θα περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για αυτά τα οποία μας παρουσιάσετε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη μεταρρύθμιση γιατί έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη σαφήνεια. Χαιρόμαστε για την νέα αυτή στρατηγική και τη νέα μέθοδο. Θεωρώ ότι προσθέτει αξιοπιστία, προβλεψιμότητα, αυτό το οποίο θέλουν και περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, ακόμη σημαντικότερο είναι ότι θα έχουμε ως πρώτο κεφάλαιο το σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος ε, δικαίου για να μπορέσει μια χώρα να ενταχθεί. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς. Αυτό το οποίο είναι επίσης ε, σημαντικό και το λέει και το όνομα μας, το Renew Europe, είναι ακριβώς ε, να δούμε την μεταρρύθμιση της Ευρώπης. Θέλουμε ε, να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να ενταχθούν βεβαίως, να υπάρξει μια πλήρης ε, ολοκλήρωση και βεβαίως θα υπάρξει και η διάσκεψη για την Ευρώπη αλλά αυτό αφορά και εσάς. Θέλω λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα. Πώς θα επηρεάσει την ε, μέθοδο με την οποία κάνετε τις ε, συνομιλίες με τις χώρες. Αυτό θα ήθελα να μου διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, για την ομάδα ID δεν έχω λάβει κάποιο αίτημα. Είστε από την ομάδα ID. Θέλετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ θέλω να καταλάβω πώς συγκεκριμένα σκέφτεστε να διαρθρώστε την ε, εγγύηση αυτή για το κράτος δικαίου σε αυτές τις ε, χώρες. Υπάρχει ένα πραγματικό δηλαδή κράτος δικαίου το οποίο θα λειτουργεί ως ε, ένα κράτος ευρωπαϊκό και σύγχρονο αλλά η μέθοδος δεν είναι σαφής. Πώς ακριβώς θα βοηθήσετε τις χώρες σε αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ για τους ε, πράσινους. Ε, η κυρία Φων Κράμον Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της πρότασης, την οποία χαιρετίζουμε και εμείς, καθώς ευθυγραμμίζεται και με τη δέσμευση της Θεσσαλονίκης και ε, ενισχύει την προσέγγιση βάση αξιών. Επίσης, χαιρετίζουμε και αυτή την ομαδοποίηση των ε, θεματικών κατηγοριών. κάτι που θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να επιβραβεύσουμε την ταχύτητα και να γίνεται αυτό με πιο δυναμικό τρόπο, ώστε να μπορούν οι χώρες αυτές να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν και πρόσβαση στις πληροφορίες και να λαμβάνουν και παρατηρήσεις από εμάς. Επίσης, θέλουμε να ε, σας χαιρετήσουμε για την ε, ευελιξία που επιδεικνύεται και την επιτάχυνση των διαδικασιών με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Όμως, υπάρχει ένα σημείο που μας ε, ανησυχεί όσον αφορά την αναθεώρηση της ε, μεθοδολογίας, που είναι η συνεισφορά των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας να υπάρχει μια πιο πολιτικοποιημένη ε, διαδικασία, να παράγονται δηλαδή αυτά τα κεντρικά δεδομένα με πολιτικοποιημένο και συγκεντρωτικό τρόπο. Θεωρούμε ότι οι εμπειρογνώμονες κομισιών θα πρέπει να είναι εκείνοι που θα συλλέγουν αυτά τα βασικά δεδομένα και όχι τα, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που ενδεχομένως να επηρεάζονται και από πολιτικά συμφέροντα. Επίσης, θα θέλαμε το κοσυφοπαίδιο να αναγνωριστεί το συντομότερο δυνατό. Εσείς μιλήσατε για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ ε, Σερβίας και Κωσόβου. Για μας στόχος είναι η πλήρης αναγνώριση. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει ένα πακέτο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής ε, τον Μάιο, οπότε θέλουμε από την πλευρά σας να προωθήσετε ένα τέτοιο πακέτο. Ευχαριστώ η Άννα Φωτίγκα για το ECR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτήν την ανακοίνωση για την διεύρυνση. Πάρα πολύ σημαντική λαμβάνει υπόψη την αντίδρασή μας σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου θεωρώ ότι με τις ε, προτάσεις αυτές ε, που έχουν παρουσιαστεί συνδυάζεται όλα όσα είχαμε ήδη πει, την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την διεύρυνση ξεκάθαρα όμως ε, και ξεκάθαρα και για τους εταίρους μας τους επιτρέπεται έτσι να αξιολογήσουν ε, την διαδικασία και για πιθανούς ε, άλλους υποψηφίους από την ίδια περιοχή που ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Καλώς όριζω το ότι τονίζεται τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης και βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει μια νέα δυναμική στην ε, διαδικασία και είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει η πιθανότητα να κλείνουν κεφάλαια. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι, δέσμη και αυτό είναι θετικό. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ σε αυτήν την πρόταση, το καλύτερο θα έλεγα, είναι τα θετικά μηνύματα. Και χρειαζόμαστε θετικά μηνύματα. ειδικά στις χώρες της ε, γειτονίας, στην διεθνή κοινότητα και τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν, ότι η διαδικασία αυτή είναι εφικτή, δυνατή και μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Το ερώτημά μου αφορά την αντίδραση της ε, Βορείου Μακεδονίας ε, και της Αλβανίας και την αξιολόγηση της αντίδρασης αυτής. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος από την ΚΟΕ τον λόγο. Α, υπάρχει. Συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση. Θεωρούμε ότι οι λαοί έχουν το απόλυτο δικαίωμα να ψάχνουν και να καθορίζουν όπως νομίζουν καλύτερα το μέλλον τους. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να κοροϊδεύουμε τους λαούς. Θέλω να μου απαντήσετε τι έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από κάποιους μήνες όταν η, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κάποιες χώρες μέλη της Ένωσης αρνήθηκαν στη Μακεδονία και στην Αλβανία το δικαίωμα της συνέχισης της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον δώσατε πάρα πολύ σημασία στην έννοια της μεθοδολογίας, πώς θα προσεγγίσουμε αυτές τις χώρες για να καταστούν κράτη-μέλη σε κάποια στιγμή. Αποφύγατε την ουσία και η ουσία για μα είναι ότι οι ακολουθούμενε πολιτικέ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν διασφαλίζουν τα οράματα και τι προσδοκίε αυτών των λαών. Ζητάτε τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποδώσατε ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Είσαστε έτοιμος να δώσετε ρόλο και ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια τη διαπραγματεύση με αυτέ τι χώρε. Ευχαριστώ. Okay, Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και θα ζητούσα από τον Επίτροπο να απαντήσει σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορεί. Ευχαριστώ. Καταρχήν έλαβα αρκετές ερωτήσεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην πολιτική καθοδήγηση αυτής της διαδικασίας. Ήδη συμβάλλει αρκετά. Και αν δείτε το έγγραφο και διαβάσετε τον έλεγχο της πρόοδου, τον έλεγχο της εφαρμογής και της υλοποίησης, διαπιστώνετε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναμίξουμε τους διάφορους θεσμικούς παράγοντες στις ε, Συμφωνίες Σύνδεσης, στο Συμφούλιο Σύνδεσης, στην Επιτροπή Σύνδεσης, και τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές σύνδεσης. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους θεσμικούς φορείς ε, περισσότερο και πιο αποτελεσματικά για να ελέγχουμε το βαθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Θέλουμε να ελέγχουμε την κατάσταση επιτόπου. Και επίσης οι επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια των χωρών ε, θα είναι σημαντικές, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του έργου το επιτελούν οι βουλές, οι εθνικές βουλές. Και προσβλέπω στην υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να με βοηθήσετε και να μου δώσετε να μου κάνετε μια αξιολόγηση των επαφών που θα έχετε με τα κοινοβούλια των χωρών και να μου πείτε πώς βλέπετε τις μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Και επίσης θα ήθελα εσείς να διαβιβάζετε κάποια μηνύματα προς τα εθνικά κοινοβούλια όταν απαιτούνται ευαίσθητες μεταρρυθμίσεις μερικές φορές ακόμη και με συνταγματικές αναθεωρήσεις. Οπότε υπολογίζω πολύ στη βοήθειά σας και νομίζω ότι θα είστε πολύ σημαντικός παράγοντας στη νέα μεθοδολογία, την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης. Κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και αναφερθήκατε και στην, ε, στο ανακοινωθέν τύπο που εξέδωσε. Πολύ γρήγορα κυκλοφορούν τα νέα. Λοιπόν, η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήδη έχουν ξεκινήσει ενταξιακέ διαπραγματεύσεις. Οπότε θα είναι δύσκολο να αλλάξουμε τους κανόνες όσο διαρκεί το παιχνίδι. Ούτε ήταν πρόθεσή μας αυτή. Πιστεύουμε πάντω ότι με την αναθεωρημένη μεθοδολογία θα καταστήσουμε πιο δυναμική και την ε, δική του ενταξιακή διαδικασία. Και υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν. Και θα σα δώσω το ίδιο παράδειγμα που έδωσα και στη συνέντευξη τύπου το οικονομικό σκέλος δηλαδή των διαπραγματεύσεων. Αν οι δύο χώρες θέλουν να επιταχύνουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα των θεματικών ενωτήτων, αυτά τα ομοδοποιημένα κεφάλαια για να το κάνουν. Και θα μπορούσαν να, να ενταχθούν σε αυτό το συγκεκριμένο, να κάνουν opt-in για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να χρησιμοποιήσουν τον νέο σύστημα των clusters, των θεματικών ενωτήτων και να χρησιμοποιήσουν την αναθεωρημένη μεθοδολογία σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Υποσχεθήκαμε να έχουμε ως χρονοδιάγραμμα το ένα έτος και αυτή είναι μια πολιτική προσφορά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας ή τη στιγμή της έναρξης της θεματικής ενότητας, θα ξεκινήσουμε ταυτόχρονα διαπραγματεύσεις για όλα τα συναφή κεφάλαια. Και εκεί οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων δεν θα αφορούν οι διαπραγματεύσεις σε κρεμές νομοθετικό έργο, αλλά την πραγματική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Οπότε αν υπάρχει βούληση για αποτελεσματική συμμετοχή των υποψηφίων χωρών, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά αυτή είναι η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξαρτηθεί φυσικά από το βαθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. από πλευράς υποψηφίων για ένταξη χωρών. Τώρα, η συμμετοχή, η συμβολή των κρατών μελών και γιατί είναι σημαντική αυτή. Από ό,τι έχω καταλάβει από τις επαφές που είχα, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται παρόμοια αξιολόγηση των ε, εξελίξεων επιτόπου. Και επειδή δεν υπάρχει αυτό το συντέριασμα, υπάρχει κάποια αντιστοιχία. Ε, γι' αυτό πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν στην ε, έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και θα έχουμε θέλουμε να αποφεύγουμε κάποιες εκπλήξεις τη τελευταία στιγμή στην αξιολόγηση. Θέλουμε να τις αποφύγουμε και να έχουμε κοινή αντίληψη για το τι συμβαίνει επί τόπου. Να μην υπάρχουν αντιστοιχίες ή παρερμηνίες από τα κράτη-μέλη. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, για να αποφύγουμε τέτοια αναντιστοιχεία και ε, κακές εκπλήξεις τελευταίας στιγμής, χρειάζεται συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών και των υποψηφίων για ένταξη χωρών. Επίσης, πώς θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να κλείσουμε και κάποια κεφάλαια. Αυτό είναι και προτεραιότητά μας και αναφέρεται στο έγγραφο της αναθεωρημένης μεθοδολογίας ότι θα πρέπει να συντμίσουμε τη μεθοδολογία που έχουμε τώρα και που εκτείνει τις διαπραγματεύσεις 6 με 8 χρόνια για τα μονομενα κεφάλαια. Σε 6 με 8 χρόνια μια χώρα έχει συνήθως δύο διαφορετικές κυβερνήσεις που αναλάσσονται. Οπότε, αν θέλουμε πραγματικά να παγιώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να κλείνουμε ταχύτερα τα κεφάλαια. Για να εδραιώνουμε τις μεταρρυθμίσεις και να έχουμε και πρόοδο στην εφαρμογή τους. Αντί να χρονοτριβούμε στα νομοθετικά βήματά τους. Τώρα, τι άλλαξε από τον Οκτώβριο. Έχουμε εκτενέστατες διαβουλεύσεις και με τα κράτη-μέλη, όχι μόνο αυτά που έχουν ανησυχήσει, που είχαν ανησυχίες και αμφιβολίες. Έχουμε επαφές με όλα τα κράτη-μέλη και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ταυτόχρονα, για να αντιληφθώ ποια είναι τα αίτια των προβλημάτων. Και τα αίτια θα πρέπει να εντοπίσουμε, τα βασικά αίτια, για να υπερκεράσουμε τις δυσκολίες της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τις δύο συγκεκριμένες χώρες. Αυτά. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Έχουμε, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, έχουμε ε, λίγο χρόνο για να κάνουμε άλλο ένα γύρο ερωτήσεων. 10 προτείνει ο Επίτροπος, 15 του αντιπροτείνει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερου συναδέλφου. Ένα λεπτό στον καθένα. Από την κυρία, η κυρία Ζόφκο από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Χαιρετίζουμε τη νέα μεθοδολογία. Είναι πολύ καλά τα νέα, ε, ιδίω για την Κροατία που είναι στα εξωτερικά σύνορα τη ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 100.000 Βόσνοι έχουν ε, κροατικό διαβατήριο και μα ανησυχεί πολύ η κατάσταση των πολιτών αυτών από την άλλη πλευρά των συνόρων. Αυτή η νέα μεθοδολογία μα δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τι προσπάθειέ μα για την διασφάλιση τη ειρήνη στην περιοχή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται περισσότερο χώρο ε, ώστε να καταθέτουν την άποψή του τα κράτη-μέλη στη νέα μεθοδολογία, που μέχρι τώρα ήταν πολύ ε, στα χέρια της Κομισιόν. Οπότε στο μέλλον περιμένουμε ε, μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου επίσης και χαιρετίζουμε αυτήν τη νέα προσέγγιση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Κιούτσουκ που είναι εισηγητής μας για τη Βόρεια Μακεδονία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίασή σας εδώ και για την προετοιμασία αυτής της νέας ε, μεθοδολογίας που νομίζω ότι θα αλλάξει την πραγματικότητα, θα δώσει περισσότερο δυναμισμό στη διαδικασία και θα μας οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή. Έχω κάποιες ερωτήσεις και ε, ανέφερε ήδη η συνάδελφος ε, Άννα Φωτίγκα ότι ήδη έχουμε ε, λάβει κάποια θετικά μηνύματα από το έγγραφο. Θέλουμε όμως και θετικά αποτελέσματα για, τον, για την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία από τη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ. Είπατε για τις ε, εκπλήξεις τελευταίας στιγμής. Πράγματι, τέτοιες ε, ε, εκπλήξεις είχαμε τον Οκτώβριο. Μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Εγώ θεωρώ πως όχι. Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα υπάρξει μια δεύτερη αποτυχία. Και τρίτο ερώτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία. Χαιρετίζουμε αυτή την ε, κατηγοροποίηση σε θεματικές ενότητες. Όμως τι θα γίνει με την ταχύτητα. Μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία, να το εγγυηθείτε αυτό ε, μετατρέποντας τους, ε, τις κατηγορίες ε, ε, διαπραγμάτευσης σε θεματικές ενότητες. Ευχαριστώ. Για το ID ο κύριος Κορόπο. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επιτρέπο. για το θέμα της διεύρυνσης η οποία αποκτά μία νέα όθηση θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό αλλά και για την ε, Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η νέα μεθοδολογία. Ε, δίνεται το βάρος στην οικονομία και στο κράτος δικαίου. Εν τω μεταξύ, οι χώρες οι οποίες είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν τεράστιες θυσίες ε, στο θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα πρέπει να αφορά και τις χώρες που αποφασίζουν να ενταχθούν, γιατί αν είναι να στηρίξουν τις χώρες οι οποίες είναι πίσω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με μία μέτρηση, 16 εργοστάσια ηλεκτρισμού στα κεντρικά Βαλκάνια εκλείουν ε, περισσότερες εκπομπές από 250 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ιδιαίτερα αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Αλφε για τους ε, πράσινους ε, ο σχεδόν ηγητής για την Τουρκία Λαγκοντίνσκι. Α, με συγχωρείτε, κυρία Στρίκ. Ευχαριστώ. Όπω είπε ήδη και ο συναλφός εμείς υποστηρίζουμε την προσέγγιση αυτή με τις δέσμες και την ευελιξία που δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει υποψήφιες χώρες την ε, διαδικασία. Όμως το πιο καινοτόμο στοιχείο βεβαίως είναι μια απόφαση να ανταστραφούν, να ανταστραφούν με συγχωρείτε διαπραγματεύσεις. Και λέει ότι σε σοβαρές περιπτώσεις η Κομισιόν μπορεί να κάνει μια πρόταση μέσω απλοποιημένης διαδικασίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό και επίσης η ψηφοφορία είναι με ειδική πλειοψηφία για να αντιστραφεί η διαδικασία. Γιατί δεν βλέπετε εδώ πέρα τον κίνδυνο ε, πολιτικής αυθαιρεσίας αλλά και της ανασφάλειας ε, που την συνοδεύει αυτήν. Αλλά και νομικά μιλώντας τώρα έχουμε ομοφωνία ε, όσον αφορά τις αποφάσεις για να προχωρήσουμε προς τα μπρος, αλλά ειδική πλειοψηφία για την αντιστροφή της εργασίας. Είναι λογικό αυτό. Σας ευχαριστώ. Εισηγητής για τη Σερβία, κύριος Μπίλτσεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα στην ανακοίνωσή σας και ελπίζω έτσι να τονιστεί η γενικότερη πολιτική προσήλωση στην ε, διεύρυνση φέτος, ε, καθώς πρέπει να προχωρήσουμε στην διαδικασία της διεύρυνσης και καλωσορίζω τη νέα μεθοδολογία. Επίσης, είναι σημαντικό να επικοινωνούμε όχι μόνο εδώ αλλά και με τους εταίρους μας στην περιοχή ε, χαίρομαι που θα πάτε τις επόμενες ημέρες σε Σερβία και Μαυροβούνιο. Επίσης θα πρέπει να ενταθεί η διαδικασία σε όλα τα μέτωπα και θα ήθελα εδώ πέρα να υπενθυμίσω την απόφαση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που ζητάει ρητά την εμπλοκή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θεωρώ ότι πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη όταν μιλάμε για το πώς θα επικοινωνήσουμε καλύτερα στα θέματα αυτά του επόμενου μήνε. Έχω μία ερώτηση. που βλέπετε στη νέα μεθοδολογία τον χώρο για την συμφιλίωση. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, είναι ιστορικό. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους τελευταίους τέσσερις πρώτα, η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε ε, και για την παρουσίασή σας. Όλοι εδώ συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αξιόπιστη και βέβαια αυτό αφορά τα πάντα Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πενεταίο το ότι ήρθατε ε, με την, και φέρατε αυτή τη νέα μεθοδολογία την οποία βρισκώ αιτιολογημένη και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι έχει στόχο να οικοδομήσει περισσότερη εμπιστοσύνη. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι σαφής ο στόχος να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία το συντομότερο δυνατόν, ίσως ήδη τον Μάρτιο. Το ερώτημα είναι πώς ε, το αξιολογείτε ε, και πώς θεωρείτε ότι θα το δουν οι χώρες ε, Χάρηκα ότι για το ότι είπατε ότι υπάρχει πλέον η επιλογή opt-in για τις χώρες οι οποίες είναι πιο προχωρημένες. Αλλά οι ίδιες πώς το βλέπουν. Ευχαριστώ κύριε Λαγκοντίνσκι. Ευχαριστώ σύντομα. Τι σημαίνει αυτό για τις άλλες υποψήφιες χώρες, ε, ειδικά την Τουρκία. Θα είναι μια ειδική περίπτωση για τα Δυτικά Βαλκάνια και αν ναι πώς θα το εξηγήσετε αυτό ε, στους ε, Τούρκους εταίρους. Σας ευχαριστώ. Και τελευταίοι δύο, Κουμπίλιος και Μάντελ. Ευχαριστώ. Η αναθεωρημένη μεθοδολογία είναι πολύ σημαντική και σίγουρα έχει πολλά θετικά. Εγώ έχω μια πιο γενική ερώτηση. Μιλούμε για την προβλεψιμότητα. Πολύ σημαντικό θέμα προβλεψιμότητα για τις υποψήφιες χώρες που θα πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις να γίνει αντικειμενική αξιολόγησή τους, αλλά προβλεψιμότητα θα πρέπει να υπάρχει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ε, για τέτοιες διαδικασίες ε, ειδική πλειοψηφία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, για το κλείσιμο κεφαλαίων, για την αντιστρεψιμότητα των διαπραγματεύσεων, γιατί θα θέλουμε κι εμείς ε, προβλεψιμότητα, όχι να μπορεί μια χώρα για ιστορικούς ή άλλους λόγους να μπλοκάρει τη διεύρυνση ή την ένταξη και ξαφνικά να παγώνει η διαδικασία λόγω μιας χώρας. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ε, ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Ο Λούκας Μάντελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πραγματικά α, ξέρουμε προς, ε, ποιος σας έβαλε αυτό το επιπλέον έργο γιατί δεν θα έπρεπε να είχαμε μπλοκάρει ε, οι διαπραγματεύσει για τι δύο χώρε και θα πρέπει να ξεκινήσουν και να απεμπλακούν και πριν την Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ. Χαίρομαι που η δημοκρατία, το κράτο δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα καλύπτονται στη νέα μεθοδολογία. Αυτό που μου λείπει όμω είναι το συνέστημα, είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή και η αντίληψή μα ότι ε, ο Σέρβο ή ο κάτοικο του Κωσυφοπεδίου είναι το ίδιο Ευρωπαίο με έναν Πολωνό, Γάλλο ή Αυστριακό. Αυτό λείπει, αυτό το, αυτή η αίσθηση λείπει και από τον κόσμο στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό το αίσθημα θα επιδεινώνεται όσο παρατείνονται οι διαπραγματεύσεις, η περίοδος για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Και η Ναταλή του Ουαζό, η τελευταία ομιλήτρια. Χαιρετίζω το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να ε, ξεφύγει από τη γραφειοκρατία η διαδικασία της διεύρυνσης γιατί η απόφαση διεύρυνσης είναι πολιτική η απόφαση και θα πρέπει να την αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποψήφιες χώρες. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται να είναι προβλέψιμη, σαφής και να προβλέπει ανάληψη ευθυνών από όλε τι πλευρέ. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Επίση, αν γίνεται πρόοδο, να λαμβάνεται υπόψη. Και αν υπάρχει οπισθοδρόμηση, επίση θα πρέπει να έχει συνέπειε. Χαίρομαι που δίνεται έμφαση στο κράτο δικαίου σε όλη την πορεία την ενταξιακή. Γιατί το κράτος δικαίου δεν είναι μόνο ένα κουτάκι που σημειώνουμε σε ένα πακέτο. Έχουμε πολλά, πολλές φιλελεύθερες δημοκρατίες ε, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε και άλλες. Επίσης, ε, δεν θέλουμε μία απλώς ε, ανακοίνωση δηλώσεων και βούλησης. Μας ενδιαφέρει η πραγματικότητα επιτόπου. Και για να διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να μεταρρυθμιστεί. Δεν μπορούμε να υποδεχόμαστε νέα μέλη σε ένα κατάστατο σπίτι. Θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στις δράσεις και στα έργα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μπορείτε να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις θέλετε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τέθηκε ένα ερώτημα για το πώς μπορώ να εγγυηθώ εγώ ε, το θετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να ζητήσω την υποστήριξη και τη βοήθειά σας για να τα καταφέρουμε μαζί. Θα είναι μια κοινή διαδικασία που θα εμπλέκει το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και βεβαίως ε, και εμένα, αλλά δεν είναι προσωπική μου υπόθεση, ε, ούτε ε, μπορώ εγώ μόνος μου να τα καταφέρω. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση σε όλους εσάς, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από τη Σύνοδο Κορυφή ε, του Ζάγκρεπ. Ποιο θα είναι το κόστο αποτυχία. Θα είναι εξαιρετικά υψηλό. Ε, έχουμε ήδη αποτύχει τρει φορέ. Είναι η τέταρτη φορά ε, και νομίζω ότι θα είναι και η τελική. Για την τελευταία φορά χάσαμε μια κυβέρνηση λόγω της αποτυχία μας. Αυτή τη φορά δεν θέλω να αποτύχουμε. Δεν θέλω να διατρέξουμε αυτόν τον κίνδυνο της αποτυχίας. Γι' αυτό και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Όσον αφορά την ταχύτητα, αυτή δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εμεί είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε τα πράγματα. Αν οι χώρε οι υποψήφιες προς ένταξη είναι επίση ε, έτοιμες να επιταχύνουν. Θα τι βοηθήσουμε αν είναι έτοιμε, αλλά δεν μπορούμε να τι βοηθήσουμε αν δεν είναι και εκείνες διατεθειμένε να επιταχύνουν. Για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και την κλιματική αλλαγή και τα σχετικά ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς θα είναι κρίσιμη σημασία η σύνοδος κορυφής του Ζάγκρεπ. Όσον αφορά της, ε, την ανάπτυξη και την οικονομία είναι και αυτά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, να τα αντιμετωπίσουν. Οι οικονομικές δυνατότητες βεβαίως είναι πολύ πιο περιορισμένες από τις δικές μας, οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε πρώτα εκείνα τα στοιχεία της Πράσινης Συμφωνίας τα οποία μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η, αποδοτικο... ενεργειακή αποδοτικότητα, η χρήση της κυκλικής οικονομίας κτλ και μπορούμε ήδη από τώρα να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές πριν από την ένταξη, ώστε όταν θα είναι πλέον μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη δουλειά μας. Είχα και ένα ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η αρχή της αντιστρεψιμότητας. Ποιες πλειοψηφίες και ποιοι μηχανισμοί θα προβλέπονται. Είναι λίγο νομικά αυτά τα θέματα. Ναι, είναι πράγματι. Ε, είναι, και, είναι και νόμιμες αυτές οι προτάσεις, ε, αλλιώς δεν θα τις είχαμε υποβάλει. Η αρχή της ε, αντίστροφης ε, ενισχυμένης πλειοψηφίας ε, είναι ε, μια τάση η οποία ενισχύεται σε διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, το TUPAC, το, το Sixpack, Frontex. Εκεί υπάρχει αυτή η αρχή και έχει εφαρμοστεί. Το σκεπτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις με την Σερβία και το Μαυροβούνιο είτε οι Κομισιόν είτε το 1 τρίτο των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν να υπάρξει αντιστροφή. Αναστολή ε, των διαπραγματεύσεων σε ένα κεφάλαιο ή και επανέναρξη διαπραγματεύσεων σε κάποιο κεφάλαιο που έχει κλείσει. Αυτοί θα είναι οι τρεις πυλώνες όπου το Συμβούλιο ε, θα έχει λόγο και όπου θα υπάρχει ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή ε, γίνεται η ψηφοφορία με ενισχυμένη πλειοψηφία. Χρειάζεται λοιπόν ενισχυμένη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή για να ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο. Αυτό που προτείνουμε τώρα είναι ότι μόνο η Κομισιόν θα μπορεί να έχει την πρωτοβουλία υποβολή μια τέτοια πρόταση. Τα κράτη-μέλη μπορούν ε, αιτιολογημένα να υποβάλουν προτάσεις προς την Κομισιόν για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, αλλά θα εξαρτάται από την Κομισιόν. Αν η Κομισιόν όμως υποβάλει μια τέτοια πρόταση, τότε θα είναι αντίστροφη ενισχυμένη πλειοψηφία θα απαραίτητη για να μπλοκαριστεί κάτι τέτοιο στο Συμβούλιο. Αυτό ε, μας δίνει ιδιαίτερη δύναμη στην όλη διαδικασία, ώστε όταν θα βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα, ελλείψεις, τότε θα μπορούμε να αναλαμβάνουμε ταχαίως δράση αποτελεσματικά και με σαφή τρόπο. Άπαξ λοιπόν και θα έχει ανακοινωθεί μια τέτοια πρωτοβουλία στην, ε, ε, προς μια χώρα, θεωρούμε ότι θα αυξήσει και την προθυμία ε, να αλλάξει τη στάση της, η χώρα αυτή, κάτι που θα μας δώσει περισσότερη δύναμη ε, ώστε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Περιφερειακή συνεργασία. Στη μεθοδολογία βλέπουμε ότι έχουμε ενισχύσει την συνεργασία σε διάφορους τομείς, χωρίς βεβαίως να, αν δεν αν, αντιμετωπιστούν οι διμερείς συγκρούσεις στην περιοχή, βεβαίως δεν μπορεί να προχωρήσει η ένταξη. Και μέσω τη στρατηγική του Ζάγκρεπ θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών, διότι σκοπός μας είναι όλο, το, οικονομικό, το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης να αφορά όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, όχι μόνο τις χώρες με τις οποίε έχουμε διαπραγματεύσει, και για το Κόσοβο δηλαδή και για τη Βοσνία Ζεγοβίνη πώς, ποια ήταν η υποδοχή ε, στις χώρες που έχουν επιδείξει επιφυλακτική στάση. Ελπίζω να είναι θετική. Θα δω και στον τύπο, από εδώ ε, θα φύγω και θα πάω στο Συμβούλιο, θα δω ε, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Πώς, ποια ήταν η υποδοχή στις ίδιες τις χώρες. Εγώ όταν επισκέφτηκα τις, δύο, ε, τις χώρες αυτές μου είπαν ότι είναι ανοιχτές και ότι είναι διατεθειμένες να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε από εμά περιμένουν στην πραγματικότητα. Όταν τους εξηγώ ε, τα σχέδιά μας, ε, αυτό με παροτρύνουν να κάνω. ότι συνεχίστε, ε, προχωράμε, είμαστε κι εμείς εδώ και θα υπάρξει συνεργασία. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Τουρκία. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι αν κοιτάξετε τη μεθοδολογία, στον τίτλο Μάλιστα θα δείτε ότι η μεθοδολογία αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Και τέλος, για το συνέστημα, ε, συμφωνώ μαζί σας, τα συναισθήματα μπορούν να είναι ωφέλιμα. Όμως το τελευταίο διάστημα ήταν τόσο φορτισμένα τα συναισθήματα που εγώ να σας πω την αλήθεια προσπάθησα κάπως να καθησυχάσω την ένταση των συναισθημάτων και να ξαναδώσω ουσία στη διαδικασία για να μπορέσουμε να την ξαναξεκινήσουμε. Και πράγματι έχετε δίκιο. Είναι όλοι Ευρωπαίοι, όπως και εμείς. Γι' αυτό και το Ζάγκρεπ θα ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να τις φέρουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο κοντά σε εμά από ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Συνάδελφοι, θα κλείσουμε σε ένα λεπτό. Απλώς να πω ότι θα ε, πάρουμε θέση για, απέναντι στην πρόταση αυτή της, ε, ε, τη νέα πρόταση της Κομισιόν εν ώψη της ε, συνόδου του Ζάγκρεπ τον Μάιο. Σας ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας, για τις απαντήσεις σας. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα που θα ήθελε κάποιος να θέσει, κηρύσω τη λήξη της σημερινής μας συνεδρίασης. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.